συνειδρίασης στην οποία μόλις αναφέρθηκα. Το πρώτο σημείο που έχουμε στην ε, ημερήσια διάταξη για το απόγευμα είναι μια προφορική ερώτηση ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ε, το θέμα της επανεγκατάστασης. Θα δώσουμε λοιπόν το